Καλημέρα σας. Λοιπόν, να μην περιμένουμε άλλο, ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία. Εγώ έχω τον κωδικό μου, έχω την κάρτα μου, τα έχουμε όλα. Ε, σήμερα έχει και απεργία από ό,τι κατάλαβα. Ε, έχει απεργία όσων είναι υπεύθυνοι για τη θέρμανση. Α, και για όσους είναι υπεύθυνους για τον καφέ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Έχει καφέ εδώ, έχει καφέ πίσω σας. Αν θέλετε μπορείτε να, να πάρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σημείο 7. Not my It's o'clock and we vote. So we start with the voting. Ξεκινούμε λοιπόν. Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Μπόρις και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε. Παρακαλώ, ποιο τρέχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι η οδηγία είναι πολύ σημαντική. Και για πρώτη φορά ε, την αναθεωρούμε μετά από τρία χρόνια για να δούμε πώ λειτουργεί. Ουσιαστικά εξασφαλίσει την προστασία τη εσωτερική αγορά και των καταναλωτών, περισσότερο δε των νέων από την υπερβολική διαφήμιση. Ταυτόχρονα όμω ε, προβάλλει και προωθεί την ελευθεροτυπία και καταπολεμά κάθε μορφή διάκριση μεταξύ των καταναλωτών. Νομίζω ότι λειτουργεί ε, η οδηγία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του και όλε τι από όλε τι πολιτικέ ομάδε για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Και τη Στεφανή Βιωσολή θέλω να ευχαριστήσω, τον Κάσα του, γιατί εργάστηκαν πολύ σκληρά. Ελπίζω και η ψηφοφορία να είναι θετική, να είναι επιτυχημένη, γιατί έχουμε άλλα ε, τρία χρόνια στα οποία θα δούμε και τη λειτουργία αυτής της οδείας και ίσως ε, εισαγάγουμε μετά από τρία χρόνια κάποιες τροποποίησεις, κάποιες βελτιώσεις. Εν γένει όμως νομίζω ότι είναι καλή για τα μέσα μαζική ενημέρωση χρειάζονται ρυθμίσει στην Ευρώπη. Θετικά πάντως ε, όλα τα βλέπω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά το χέρι σα, γιατί δεν βλέπω μέσα σε, αυτό το, σε αυτή την αίθουσα. Ή θα ψηφίσουμε τα πάντα ηλεκτρονικά, ή θα κάνετε λιγάκι γυμναστική το πρωί. Σήμερα θα σηκώνετε το χεράκι σας ψηλά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Χωριστή ψηφοφορία. Ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το 55 το 55 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά okay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 Είσαστε κατά ή είσαστε υπέρ. Κατά είσαστε. Μάλιστα. Ωραία. Άρα 8 ε, με 12 απορρίπτεται. 56 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τριαβολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 67. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Vote is closed. ψηφοφορία. Zu 12. 19 ψηφίσαντε. 8 υπέρ, 12 κατά απορρίπτεται. 8 με 13 λοιπόν. Απορρίπτεται με πάση περιπτώσει. Ε, η 68 είναι παρόμοια. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ. Υπέρ. Για την 71. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. 71. Vote is closed ψηφοφορία. 16 17 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 88. Vote closed. Πέρας. 14 υπέρ 10 κατά. Μην, σας μετράω, μην ανησυχείτε, σας μετράω. 15 με 10. Εγκρίνεται λοιπόν. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 92. Όχι. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 και λίμπε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 116. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 9 προς 15, 10 προς 15. Απορρίπτεται λοιπόν. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε για τη 10 λέει η πρόεδρος. Πέρας. Α, ναι, έχετε δίκιο. Δεν έκανα λάθος. 11. Δεν ξέρω, λέει πρόεδρο. Την 11, την 11. Η 10 εγκρίθηκε. Και η 11 εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συγγνώμη γι' αυτό. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές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 Πέρας ψηφοφορίας. 7 προς 16, άρα 8 προς 16. Κύριε Χάνιμπαλ, τι ψηφίζετε υπέρ. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Όχι, εγκρίνεται. 26 υπέρ. Συγγνώμη. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές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 απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στη Λίμπε. Λίμπε 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τις τέσσερις επόμενες μαζί μπορούμε. 7 με 11. Όχι, δεν μπορούμε. 7 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 14, ναι, 13. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε για τη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 προς 10. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν τώρα με την ηλεκτρονική κάρτα. Ποιος δεν έχει, με την κάρτα λοιπόν ψηφίζουμε την... You, can do it with your Mastercard, okay. Βάλτε Mastercard, δεν πειράζει. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία. Πέρας. Καταψήφισα, λέει ο κύριος, Βεβαίω, βεβαίως. Λοιπόν, η κυρία Χάνιμπολ τι έχει κάνει. Εσείς έχετε κάρτα, οκ. Λοιπόν, 21 προς 23, που σημαίνει φιλελεύθερη, 3, συγγνώμη, 21 προς 3, άρα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. The liberals have to show that they are close to the pirates, huh? Isn't it? No? Not this time? Okay. You can stay. We have another vote. Μην φεύγετε, Μαρίκη, γιατί έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Επαρνάμε λοιπόν στο επόμενο. Mr. and, um... Πάμε στην έκθεση Lockegaard. Which one is it? Okay. Seven. Okay. So, Mr. Lockegaard, do you have to say...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 22 ψηφίζατες, 21 ψήφοι υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε, κάνατε πολύ καλή δουλειά. So, now we come to the next... Πάμε στο επόμενο σημείο. Σημείο 9. Ναι, όχι 9. 9. Μαρή Τερές Sánchez Σμιντ όθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Εχτες κάναμε τις συναντήσεις των συντονιστών και συζητήσαμε για το θέμα αυτό, την ε, προώθηση και τον πολιτισμό και τη δημιουργία. Πρέπει να σας πω ότι εχτες από τον νέο διευθυντή του α, ε, Τμήματος Πολιτισμού με, με, με προειδοποίησε ότι αυτό το Creative Europe δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως όνομα γιατί υπάρχει στα γαλλικά ε, το ε, Europe Creative υπάρχει στη Γαλλία κάτι, υπάρχει μια τέτοια ένωση και ε, επιμένουν ότι είναι δικό τους όνομα το Creative Europe και για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς πρέπει να πληρώσουμε. Οπότε επειδή εμείς δεν θέλουμε να πληρώσουμε πρέπει να βρούμε άλλο όνομα. Οπότε σκεφτείτε αν μπορούμε να βρούμε ένα διαφορετικό όνομα για τούτο το πρόγραμμα. Ε, Ούτω ή άλλω δεν μα είχε αρέσει και από την αρχή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έκθεση πρωτοβουλία τη Μαρή Τερέζ. Και να πω ότι ε, αποφασίσαμε να γίνει και μια ακρόαση για το θέμα αυτό. Μαρή Τερέζ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Ντορί που με επιτρέπει να ε, εκφραστώ στο πλαίσιο αυτή τη πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων για την πρόθεση του τομέα της πολιτισμού και τη δημιουργία. Ε, υπάρχουν διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το θέμα. Πάντω, κατά βάση ο στόχος μας σήμερα είναι να ευνοήσουμε τη μεγέθυνση και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας. Να σας θυμίσω ότι η Κομισιόν τον περασμένο Οκτώβριο δημιούργησε έναν ανακοινοθέν για αυτό το τομέα μετά από το πράσινο βιβλίο του 2010, επί το οποίο είχαμε ψηφίσει μια έκθεση την οποία εγώ είχα την τιμή να συντάξω. Είχαμε σκεφτεί για τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν ώστε να απελευθερωθεί το δυναμικό αυτού του τομέα και φαίνεται πως το καταφέραμε διότι η ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνει πολλές από τις προτάσεις μας. Μια σύντομη υπενθύμηση, αν και δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι περνάμε κρίση. Ο στόχος μας πάντως είναι ξεκάθαρος και μάλιστα περιλαμβάνεται στον τίτλο αυτής της έκθεσης να ευνοηθεί η μεγέθηση και επασχόληση. Δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά να βρούμε συγκεκριμένες ε, ε, οδούς που μπορεί να ωφελήσουν. Ο τομέας του πολιτισμού προοδεύει παρά την κρίση και ευνοεί την λάμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω και μάλλον και εντάσσεται στους στόχους της στρατηγικής 2020, δηλαδή μεγέθυνση βιώσιμη, ευφυή και πρακτική. Τονίζουμε λοιπόν συγκεκριμένους τρόπους. Καταρχήν τις προκλήσεις. Διπλός ο στόχος να επιβεβαιώσουμε την ιδιαιτερότητα του τομέα που χαρακτηρίζεται από διφή φύση, δηλαδή πολιτιστική και οικονομική, ε, ότι επίσης ο τομέας του πολιτισμού δημιουργεί πλούτο ίσως περισσότερο από άλλους τομείς σε αυτή την φάση. Και επίσης ανοίγει κοινωνικά στον ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης έχουμε στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχουμε τις τοπικές αρχές ε, που διατηρούν το ε, πολιτιστικό πλούτο που είναι ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και βελτιώνουν την γέθνηση και την απασχόληση. Θα πρέπει επίσης να το στηρίξουμε σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, δηλαδή τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, την ανάγκη για προσαρμογή ψηφιοποίηση και την πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης που παραμένει δύσκολη. Ε, πώς θα εναρμονιστούν τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης εθνικά, περιφερειακά και τοπικά. Εδώ το πρόβλημα. Η Κομισιόν ίσως εδώ δεν προχωρά αρκετά στα μέτρα που προτείνει και ελπίζω πως η έκθεσή μας θα αποτελέσει πηγή έμπνευση. Να θυμίσω ίσως κάποια στοιχεία που δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστα γιατί διαφέρουν ανάλογα με τις μελέτες και ανάλογα με τον ορισμό του τι είναι η βιομηχανία της δημιουργίας. Μια μελέτη του 2010 λέει ότι πως αν αναθεωρήσουμε την κεντρική δημιουργική ε, βιομηχανία, δηλα... αντιπροσωπεύει το 7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, 14 εκατομμύρια θέσεις αποσχόλησης και 860 δις ε, ετήσια έσοδα. Πώς θα δείξουμε ότι αυτός ο τομέας ε, προοδεύει παρά την κρίση. Το 2000, α, μάλλον, ανάμεσα στο 8 και το 11 η επασχόληση στον τομέα αυτό ε, αντιστάθηκε περισσότερο. Ωστόσο βλέπουμε ποσοστά μεγέθυνσης διαφορετικά από τον έναν υποτομέα στον άλλον και αυτή η τάση είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί πολλοί τομεί εδώ απασχολούν περισσότερους νέους. Οι διαφορές είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. Ο τομέας του CD και του DVD έχει χάσει μεγατμήμα του τζίρου του. Η Virgin Megastore έχει απολύσει στη Γαλλία, ενώ έχουν αναδυθεί διάφορα site online επιγραμμικά. ενώ τα προϊόντα Lux πολυτελείας ε, συνεχίζουν να, να, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αύξηση του χάσματος ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Έπειτα, στρατηγικέ ε, επενδύσει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έδωσαν θεαματικά αποτελέσματα. Τα φεστιβάλ, οι πρωτοβουλίε ε, των ευρωπαϊκών πρωτευουσών πολιτισμού γεννούν πολύ σημαντικά οικονομικά ωφέλη που πολύ συχνά διπλασιάζουν κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί, για παράδειγμα όσον αφορά την αστική ανάπτυξη για τι ευρωπαϊκέ πολιτιστικέ πρωτεύουσες. Ποια είναι τα ατού αυτού του τομέα, οι θετικέ πτυχέ που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Καταρχήν η ιδιαιτερότητα που, του που, δημιουργεί, που, καθιστά μια χωριστή οικοτομία που αντιστέκεται καλύτερα στην κρίση ιδιαιτερότητες. Είμαστε μπροστά σε ένα οικονομικό οικοσύστημα πολύ ανομιογενές που αποτελείται από διάφορους φορείς διαφορετικών μεγεθών και πρέπει να ευνοήσουμε την ανάδυση μιας κοινή ταυτότητας μέσω της προσέγγισης δικτύων και χώρων διαλόγου. Για να γίνει αυτό, θυμίζω τα τεχνικά μέσα της Κομισιόν και της, ε, των κρατών Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για να φτάσουμε σε μια πιο συγκεκριμένη στατιστική εκπροσώπηση αυτού του τομέα για να μετρήσουμε ακριβώς δηλαδή τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνουμε για τη δημιουργία, για τα συστήματα, για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με κατάλληλο τρόπο. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συντονιστές που δέχτηκαν να, διοργανώσουμε μια κρόση με εμπειρογνώμονες για αυτό το σύστημα και που θα μπορούσαν να μας δώσουν ε, στοιχεία ποσοτικά. Έπειτα, αριστεί και ανταγωνιστικότητα του τομέα, της δημιουργίας και του πολιτισμού που προσφέρουν διεθνή διάσταση της Ευρωπής ε, της δημιουργικής και της πολιτιστικής. Ευνοούν νέα μοντέλα επιχειρηματικά και νέα προστιθέμενη αξία για προϊόντα και διαδικασίες που μπορούν να εντοπιστούν. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό ως προϊόντα αριστείας στο διεθνή αγορά. Και έπειτα η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, μια διεθνής διάσταση της Ευρώπης, ε, δίνει νέα όθηση στο, στον ε, διαπολιτισμικό διάλογο, όπως αυτό συντάσσεται στη διάσταση, στην ε, σύμβαση της UNESCO. Ας πάρουμε ακόμα μια φορά το παράδειγμα των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτοβουσών, που είναι εκδηλώσεις μεγάλης αξίας, που τονίζουν τον πλούτο, τη διαφορετικότητα και τις ε, ε πτυχές των, ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με την πρωτοβουλία της, του σήματος, του Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς μπορεί να δώσουμε όθηση στη συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, ε, η εξαίρεση, η περίφημη εξαίρεση πολιτιστική, οι βιομηχανίες πολυτελείας, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύουν ε, διάφορα επαγγέλματα, βιοτεχνικά και ε, πρόκειται για τα χώρους όπου μεταδίδονται οι πιο, λεπτο, πιο πολλές λεπτομέρειες για κάθε επάγγελμα, αλλά και είναι και τα φυτόρια των δημιουργικών ε, επιχειρήσεων αυτά. Εδώ μπορούμε να δούμε τους νέους τρόπους ε, διάδοσης με το πέρασμα στην ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες για τη διαδικασία παραγωγής ε, και διανομής, την πειρατεία, την πλαστογράφηση, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μέσα και να προστατεύσουμε τα, ε, τις δημιουργίες με μέσα ελαστικά και αποτελεσματικά, γιατί αντιμετωπίζουν ψηλό επίπεδο κινδύνου. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς, την έλλειψη συνεργασίας και τις νέες συμπεριφορές των καταναλωτών πώς θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Εδώ θα πρέπει να προβούμε σε προτάσεις. Ποιοι είναι οι τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να παρέμβει για να βελτιώσει το δυναμικό αυτών των τομέων, ώστε να αυξήσει το εφέ μόχλευσης για την ανάπτυξη και την ε, απασχόληση, καινοτομία και ξανά καινοτομία νέες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στον τομέα της πολυγλωσσίας, για παράδειγμα, ευνοώντας ε, τον υποτιτλισμό ή μεταγλωτισμό των ε, ταινιών ε, ενισχύοντας ε, την ολοκλήρωση ανάμεσα στις στρατηγικές και την εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και επίσης καταρτίζοντας νέους και λιγότερο νέους σε θέσεις αριστείας. Έτσι θα πρέπει να ενεργήσουμε πολλαπλασιάζοντας τις ανταλλαγές ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και τον ακαδημαϊκό. Φυσικά, στην, επιμένοντας στη δική μας νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, θα κάνουμε οικονομίες όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού, τον εργα... το εργατικό δίκαιο, αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ανάπτυξη αυτών των τομέων. Ανάπτυξη αρμοδιοτήτων, προώθηση νέων εμπορικών μοντέλων, ε, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ε, αλλά και πέρασμα προς άλλους τομείς. Η χρηματοδότηση, η πρόσβαση ε, στην στήριξη των οικονομικών φορέων, ε, οθώντας τους επενδυτές για να ευνοήσουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το δυναμικό αυτών των τομέων και τη σύνδεσή τους με άλλους κλάδους της οικονομίας. Τέλος, θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και ήδη το είπα αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι τα διευθυντικά ταμεία μπορούν και οφείλουν να κινητοποιηθούν για να στηρίξουν τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Η πολιτιστική ε, πολιτική της Ένωσης βασίζεται σε ένα δις ευρώ ενώ ε, τα ε, διευθυντικά ταμεία έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 400 δις ε, για τις επενδύσεις τους. Έτσι θα μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, η προώθηση δε αυτού του προϊόντων θα πρέπει να προωθηθεί και μέσω χαμηλότερης φορολογίας για τα πολιτιστικά αγαθά είτε με την ε, παράταση των συστημάτων ε, των εθνικών ενισχύσεων. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Σε ένα ιδιαίτερο κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει ένα μέσο όρο ανάμεσα στι ρυθμιστικέ απαιτήσει, ανταγωνισμό, κρατικέ ενισχύσει, πρόσβαση σε όλου και το δυναμικό, το οικονομικό που δεν θα πρέπει να το ε, ε, αποδυναμώσουμε ε, μόνο λόγω διαφόρων κανόνων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι ο κλάδος αυτός έχει, επηρεάζει την ανάπτυξη, ο χρόνος πιέζει γιατί ο ανταγωνισμός είναι παγκοσμίου επίπεδου. Ευχαριστώ. Ο Σαντιάγο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Μαρή Τερέζ. Μαρή Τερέζ είναι πληρέστατη εκθεσή σου και άκρο ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, το ανέφερε και εσύ, τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δείξουμε στις κυβερνήσει μας, στις περιφέρειες, ε, στους Δήμου μα, ότι γενικά Κάθε ένα ευρώ το οποίο επενδύεται στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ε, Παραδείγματο χάρη σε άλλου τομεί όπω είναι ο τουρισμό, ε, τα φεστιβάλ. Ε, το βλέπουμε. Πολλέ φορέ βλέπω εδώ να περικόπτονται οι ενισχύσει προ τα φεστιβάλ ενώ εν γίνει η διοργάνωση ενός φεστιβάλ προσελκύει κοινό, όχι μόνο τοπικό, αλλά και από άλλες περιοχές, είτε από την ίδια χώρα, είτε από το εξωτερικό. Άρα οι επενδύσεις, οι δαπάνες ε, για τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ, επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά ε, υπερπολαπλασιάζονται, νομίζω πενταπλασιάζονται, ε, γιατί έχουμε συμπληρωματικά ωφέλη στον τομέα της, του τουρισμού, των ξενοδοχείων κτλ. Άρα μπορούμε να δείξουμε στους πολιτικούς οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, κυρίως όμως και με τα οικονομικά, αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που έχει ο πολιτισμός, για να μην μιλήσουμε για την κληρονομιά που νομίζω είναι κάτι από τα σημαντικότερα στοιχεία και σημαντικότητα τους πόλους έλξης στην Ευρώπη και πρέπει να το φροντίζουμε, να διαφυλάτουμε αυτή την κληρονομιά. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον είναι δυνατόν αυτό, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε ένα είδος ε, χορηγίας ε, σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο όπως υπάρχει στην ε, Αμερική με σύγχρονους με οι οποίοι θα επενδύουν στην, στον πολιτισμό που βέβαια ενδιαφέρονται να το πράξουν διότι αλλιώς θα είναι δύσκολο. Και κάτι ακόμη, υπάρχει μια άλλη πρόταση στην Ισπανία Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται το 1% για τον πολιτισμό, δηλαδή όλα τα δημόσια έργα που γίνονται είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Από αυτά το 1% αφαιρείται και αφιερώνεται στην πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή ε, στην επένδυση ε, αγορά έργων τέχνης για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν αυτό μπαίνει στα τρέχοντα έξοδα και αν θα ήταν δυνατόν να κάνουμε μια σχετική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, με τον τόσο εντυπωσιακό προπολογισμό που έχουμε για επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1% θα μπορούσε να προορίζεται για τον πολιτισμό εν γέννη. Είναι αυτή μια πρόταση νομίζω που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Θα ήταν κάτι καινοτόμο. Ίσως κάποιοι ε, να διωθούν. Αλλά γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Danke. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ δύο πράγματα να πω. Ε, μετά από τις πρόσφατες συναντήσεις που είχα τούτη την εβδομάδα, όπου συζητήσαμε τις ε, ε εταιρείες ε, ή το, τις ομάδες συλλεκτών για την, και για τη μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει η Κομισιόν, θα το ξαναδούμε βέβαια και τις επόμενες εβδομάδες αυτό. Έχουμε και μια διάσκεψη η οποία έγινε χτες και προχτές εδώ στις Βρυξέλλες σχετικά. Και κάποιος από τις 100 χώρες είπε ότι με την ψηφιακή επανάσταση και με τις νέες ε, Δυνατότητε διανομή που έχουμε με τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, και ξέρουμε ότι πολλές πλατφόρμες το εκμεταλλεύονται, ότι η βιομηχανία που έχει να κάνει με τη διανομή περιεχομένου ή η βιομηχανία δημιουργικού ουσιαστικά αν δεν, έχει, ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εγωγούς. Ε, οπότε δεν, πρέπει να τονίσουμε τον, α, τα ωφέλη που μπορεί να υπάρχουν ε, για την βιομηχανία αυτή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς περιεχόμενο δεν μπορούμε να έχουμε τελικά κανένα αποτέλεσμα. Και επίσης, ε, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συνδέσει, ε, να το περιλάβει στην εκθεσή σου, Μαριτερέ, είναι ότι αν θέλει κανεί να επενδύσει περισσότερα στον πολιτισμό, τότε πρέπει να, έχουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση η δημιουργία απέναντι στους παραγωγούς ή άλλους που συνάπτουν συμβάσεις μαζί τους. Επομένως, μία από τις προτάσεις είναι η μεταρρύθμιση του ενοχικού δικαίου. Ακριβώ για να έχουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση οι δημιουργοί. Ίσως αυτή την ιδέα θα μπορούσαμε να την συμπεριλάβουμε με κάποιο τρόπο στην έκθεσή σου, γιατί είναι ούτως ή άλλως και ένα θέμα που εμπίπτει στα ευρύτερα πλαίσια της στρατηγική ε, και την ε, γενικότερη δημιουργία και την καλύτερη αποζημίωση των καλλιτεχνών. Χωρί μικρόφωνο η πρόεδρο. Άλλο κανείς θέλει το λόγο. Ο Μόρτεν.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 Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε όσοι είμαστε σε τούτη την αίθουσα ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε την, τον κλάδο αυτό. Βεβαίως ε, βλέπουμε ότι και η Κομισιόν ε, κινείται στην ίδια άγουσα. Η μεγάλη βεβαίως πρόκληση είναι ε, να ότι πρέπει να, ε, να επηρεάσουμε και να πείσουμε και άλλους ε, ευρωβουλευτές. Δεν έχει νόημα να καθόμαστε εδώ στην αίθουσά μας και να μιλούμε μεταξύ μας και να μην ε, πείσουμε και άλλους για τη σκοπιμότητα αυτής της ε, διαδικασίας. Οπότε πρέπει να είναι, ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο για τους ίδιους τους δημιουργούς αλλά για την Ευρώπη, για την ανάπτυξη αυτή η ιδέα να συνδεθεί ακριβώς με την πολιτική για την ε, ανάπτυξη. Επομένως, ε, καλό θα ήταν σε αυτή την έκθεση να κάνουμε ίσως κάποιες ε, σκέψεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε τον πολιτιστικό τομέα να τον προωθήσουμε, γιατί εφόσον θέλουμε να τον προωθήσουμε πρέπει να δώσουμε και κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να συμβάλλει ο καθένας που εμπλέκεται στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει και μια πολιτιστική προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι ε, λείπει και ε, ε, η ενσυνείδητη σύμπραξη και του πολιτιστικού τομέα. Ίσως θα πρέπει να θέσουμε κάποιες απαιτήσεις, ας πούμε, και προς τους δημιουργούς, γιατί και οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν με στρατηγικό τρόπο για να μπορέσει να υπάρξει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Α, συγγνώμη. Η κυρία Νίγκε είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την Επιτροπή σας για τη δουλειά που κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Πέραν ε, της ε, μεγάλης αξίας που έχει ο πολιτισμός και το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Εν συντομία, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία μιας πολιτικής βασισμένης αποδείξης, evidence-based. Και πρέπει και τα κράτη-μέλη να ευαισθητοποιηθούν. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περσινού Νοεμβρίου αναφέρεται το ζήτημα πιο ποιοτικών στατιστικών στοιχείων για τον πολιτισμό και ιδίως ό,τι αφορά τον τομέα, τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό. Γίνεται δουλειά σε επίπεδο Eurostat Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ε, που μόλι δρομολέξει και μια μελέτη για την απασχόληση στον ε, δημιουργικό πολιτιστικό τομέα και ελπίζουμε το επόμενο έτος να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατάσταση της απασχόλησης στο μέσα αυτούς. Εθνικοί λογαριασμοί για τον πολιτισμό. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη ένα τέτοιο εθνικό λογαριασμό. Τα άλλα κράτη ελπίζουμε να μιμηθούν το παράδειγμα αυτό σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση κατ' εμάς είναι το σημείο κλειδί και στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου. Και αυτό μπορούμε να το πλασάρουμε στα κράτη-μέλη, στις περιφέρειες και στις πόλεις. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της ανακοίνωσης μιλάμε για εγκάρσεις στρατηγικές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι θα δημιουργηθούν πραγματικές συγκεκριμένες ευκαιρίες για τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ένα τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το οποίο εσείς ε, είχατε την πρωτοβουλία και θέλω να σας ευχαριστήσω. οικονομία της πολιτικής ποικιλομορφίας λέγεται αυτό το πρόγραμμα. Στόχο, είναι να βρούμε καινοτόμε ιδέες σε σχέση και με τις τεχνολογίε πληροφοριών και επικοινωνιών. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και την πρόοδο αυτής της μελέτης. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλες τις ε, παρεμβάσεις. Από όλα όσα είπαμε, νομίζω ότι πράγματι ε, πρέπει να τονίσουμε το θέμα της ευαισθητοποίησης. Βέβαια, ο Μάρτεν είπε να πείσουμε και προτιμώ αυτό τον όρο. Πρέπει να πείσουμε ότι ο πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο έχει προστιθέμενη ξένα προσφέρει. Και δεν μιλάμε μόνο για τα οικονομικά και τον προπολογισμό εδώ. Βέβαια βλέπουμε πόσο σημασία έχει ο προπολογισμό ο οποίος μπορεί να διτεθεί για την παιδεία και τον πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε και στήριξη μέσω έρευνα καινοτομία και διαρθρωτικών ταμείων και από άλλα κονδύλια δηλαδή του προπολογισμού. Αλλά κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε οποιοδήποτε μέσο ε, προώθηση του πολιτιστικού δημιουργικού τομέα. Υπάρχει προστιθέμενη αξία. Απλά πρέπει να τη δείξουμε να την ε, προβάλλουμε και να προωθήσουμε και το τεράστιο δυναμικό που έχει. Επίσης πρέπει να δούμε η ανάπτυξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου, ο πολιτισμός εν γέννη, τι προσφέρει καθημερινά στους πολίτες. Εγώ πολλές φορές μιλώ και για την καλλιτεχνική πολιτιστική εκπαίδευση. Ό,τι όμως επιτρέπει την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στον πολιτισμό είναι να... Ε, στοιχείο που πρέπει να το προωθήσουμε. Υπάρχει όμως και οικονομική δυναμική από πίσω, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για πολιτισμική, ή πολιτιστική εξαίρεση, γιατί έχει αυτή αυτό το διφύ χαρακτήρα πολιτισμικό και οικονομικό. Χαίρομαι πολύ που η Eurostat αποφάσισε να αναθέσει αυτή τη μελέτη για την απασχόληση στον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο και αυτό θα μας δώσει και επιχειρήματα για να πείσουμε για τη μεγάλη σημασία του κλάδου να πείσουμε για τη μεγάλη του συνεισφορά στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ανάδειξή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Και συμφωνώ και εγώ με τη σημασία που έχει σε όλα τα επίπεδα να γίνει αυτό τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Πρέπει να πείσουμε ότι οι κλάδοι αυτοί, οι τομείς πρέπει να υποστηριχθούν. Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τον κανονισμό και κάθε φορά πρέπει να λέμε τα ταμεία, τα προγράμματα πρέπει να είναι προσβάσιμα και για όλα τα πολιτισμικά προγράμματα τη ενία. Γιατί ο στόχο των διαφορετικών ταμείων, μεταξύ άλλων, είναι και η πρόθεση τη ανταγωνιστικότητα μέσω των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο. Και πρέπει να σα πω ότι εκτό αυτών μεγάλων επιχειρήσεων στον τομέα της, ε, του ακουστών, του οπτικοακουστικού, του κινηματογράφου κτλ., υπάρχουν και πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει και πολύ μικρέ επιχειρήσει που και αυτέ συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα έχουμε λοιπόν σύντομα και ακρόαση. Και καλό είναι να συσχετίσουμε την ηθική με ε, τον πολιτισμό γιατί μπορούν και αυτοί ε, να προσφέρουν ένα λιθαράκι. Οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη οικονομία. Ίσως κάποιος να μην τα σκέφτεται σήμερα, αλλά υπάρχουν προσεγγίσεις από κάποιες επιχείρησεις προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη από σήμερα. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι η διασύνδεση με άλλου τομεί είναι πολύ σημαντική και βεβαίω πρέπει να την έχουμε πάντα υπόψη μα. Χθε το απόγευμα στου συντονιστέ αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε μία ακρόαση τον Απρίλιο και γι' αυτό ε, θα πάει λίγο προς το φθινόπωρο η γνωμοδότηση. Θα, κάνουμε το, θα έχουμε το σχέδιο ε, έκθεσης ε, τον Ιούνιο. Οπότε θα μπορέσουμε έτσι να, το να συμπεριλάβουμε μάλλον στην έκθεση αυτή ό,τι νέο προκύψει από την ακρόαση του Απριλίου. Και έτσι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβρη. Οπότε ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα γιατί το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος δεν θα το δούμε σήμερα. Ε, θα ήταν μια ανταλλαγή απόψεων ε, σήμερα, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Χίρση, αλλά η κυρία Χίρση είναι σε άλλη επιτροπή και δεν μπορεί να είναι εδώ. Οπότε τη βάλαμε για την επόμενη ε, συνεδρίασή μας. Είναι σημαντικό θέμα βεβαίως αυτό, γιατί πιστεύω ότι με αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα μπορούμε να κάνουμε πολλά για, την, για να υποστηρίξουμε τον τομέα της, ε, ε, του πολιτισμού. Ε, για σήμερα λοιπόν το μόνο που έχουμε είναι ότι ε, λήφθησαν πολύ καλές αποφάσεις από τους συντονιστές, ελπίζω να μην έχει κάποιος αντίρρηση. Όχι. διάφορα δεν έχει κανένας. Επόμενη συνεδρίαση 20 Μαρτίου στις 10 για όλη την ημέρα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος ευχαριστεί τις, τους διερμηνείς. Α, τους διερμηνείς τους χρειαζόμαστε ε, για την συνεδρίαση που έχουμε στη συνέχεια. Όποιος ε, δεν χρειάζεται να παραμείνει στην αίθουσα, ας αποχωρήσει, γιατί θα πάμε κατευθείαν ε, στο θέμα με το European Citizenship και θα δούμε τι θα κάνουμε και με το σχετικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα το συζητήσουμε τώρα. Ο κύριος Στάκουλα είναι ο εισηγητής.